12. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο 5η, 23 Ιουνίου, από τις 8.30 έως τις 13. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λίγη συνεδρίαση. Καλή σας νύχτα.